163 του κανονισμού. Και τώρα περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη. Χαιρετούμε την Επίτροπο που έμεινε εδώ μαζί μας μέχρι βαθιά νύχτα. Λοιπόν, προχωρημένη ώρα. Για την ειδική έκθεση του Μεσομελευητή για την έρευνα για που ξεκίνησε η πρωτοβουλία που ξεκινούν η ίδια πρωτοβουλία. Πόλτσακ. Έχετε το λόγο. Συνάδελφε Πόλτσακ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θέλω να πω ότι υποστήριξα την έκθεση αυτή διότι τα συμπεράσματα είναι ορθά. Έχω κάποιο σχόλιο όσον αφορά με συγκεκριμένη ψήφ ψηφοφορία που αφορούσε την ειδική προστασία των ανηλίκων και των ΛΟΑΔ. Εγώ δεν υποστήριξα αυτό το σημείο, όχι διότι πιστεύω ότι αυτές οι ομάδες δεν αξίζουν υποστήριξης και προστασίας, αλλά προσπάθησα να εφαρμόσω την άποψη κατά την οποία αν λες ότι είσαι ΛΟΑΔ δεν θα επιστραφεί στην χώρα στην, από την οποία ήρθες γιατί μπορεί να σε κακομεταχειριστούν, κακομεταχειριστούν συγγνώμη κλπ. Εγώ νομίζω ότι είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι κανείς μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι ΛΟΑΔ. Πώς θα το επαληθεύσουμε. Θεώρησα ότι δεν μπορούσα να το υπερψηφίσω αυτό. Ευχαριστώ. Πάμε στην έκθεση Καριμαντέλη για την βιώσιμη αστική κινητικότητα. Και πάντα ο κύριος Πόλτσακ έχει το λόγο. Και ο κύριος Πόλτσακ λέει. Λοιπόν, πάλι εγώ πρέπει να πω Ευχαριστώ. Δεν μπόρεσα να υπερψηφίσω αυτή την έκθεση για ε, διάφορους λόγους. Σας ακούμε, σας ακούμε, σας προσέχουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ομιλώ και θα συνεχίσω με την παρέμβασή μου. Λοιπόν, εντάξει, ξαναξεκινώ. Δεν ήμουν σε θέση να υπερψηφίσω αυτή την έκθεση και αυτό για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι η η υποστήριξη εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό υπερβαίνει τα εσκαμμένα η πρόταση ε, εκείνων που θα ήταν λογικές προτάσεις που δεν θα παραβίαζαν την αρχή της επικουρικότητας. Θα ήταν πολύ καλύτερο αν αυτά τα θέματα τα αφήναμε να ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό όχι επειδή είμαι κατά των ποδηλάτων και της χρήσης τους στις πόλεις, στα αστικά κέντρα. Ίσα ίσα δεν είναι όμως αναγκαίο να υπάρχει ρύθμιση ευρωπαϊκή ή ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα. Από την άλλη πλευρά τα έθνη, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ρυθμίζουν αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ κύριε Πολτσακ. Έχω λάβει πολλά αιτήματα επεξηγήσεων ψήφου, προφορικών επεξηγήσεων ψήφου. Επισημαίνω ότι άλλες δηλώσεις επεξηγήσεις ψήφου μπορούν να υποβληθούν γραπτός. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση όσον αφορά τις ερωτήσεις. Τα πρακτικά της, της ε, συνεδρίας.